Good afternoon. I am very surprised because... Καλησπέρα σας. Με εντυπωσιάζει ότι το πρωί στις 9 και 10 είχα πολύ λιγότερου συναδέλφους από ότι τώρα παρόντες. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο άδεια ήταν η αίθουσα mm. στην αρχή της συνεδρίασής μας σήμερα το πρωί στις 9. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας με το σημείο 13. Η επίτευξη της, ε, του στόχου 10% της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας ε, για να, ένα επαρκές ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020. Έχουμε τον συνάδελφο Πέτερ Έριξον. Και είναι μαζί μας και θέλουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. όπως γνωρίζετε, αποτελεί ένα συγκεκριμένο βήμα προς την Ενεργειακή Ένωση. 10% ε, στόχος ε, για, την, ε, για ένα σύστημα διασύνδεσης για την ηλεκτρική ενέργεια. Ρεαλιστικό στόχος για το σύνολο της Ένωσης. σημαντική συμβολή για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού. Όταν μιλάμε για ασφάλεια ανεφοδιασμού, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο βήμα, όπως στην περίπτωση του ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο με την αντίστροφη ροή. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στον ηλεκτρισμό είναι χαρακτηριστικό το εναλλασσόμενο ρεύμα στους, ε, στους, ε, στις συνδέσεις, στις διασυνδέσεις του ηλεκτρισμού, ενώ στο φυσικό αέριο δεν είναι πάντα. Ο κύριος Έριξαν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, η έκθεση αυτή και το θέμα της διασύνδεσης είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό κομμάτι της Ενεργειακής Ένωσης, διότι τα περισσότερα από όσα θέλουμε να πετύχουμε εξαρτώνται από το αν μπορούμε να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Σήμερα δεν έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά τη μέρα που θα το πετύχουμε θα καταφέρουμε ε, να πετύχουμε και πολλούς από τους άλλους στόχους μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και χαίρομαι πολύ για τη συνεργασία που είχαμε τους συναδέλφους, τους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους η συνεργασία ήταν θετική. Είχαμε πολύ χρήσιμες συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Προσπάθησα να εργαστώ με διαφανή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων πετύχαμε καλή συνένεση για τα σημαντικά θέματα. Ίσως να μην χρειαστεί και πολύ χρόνος για τους τελικούς συμβιβασμούς. Θα δούμε όμως τι θα γίνει σήμερα και θα μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Τα πιο σημαντικά θέματα η ενίσχυση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ε, το να έχει περισσότερο προσωπικό για να ε, μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του, να υπάρχει ε, ένας μηχανισμός ελέγχου που να εποπτεύει τα εθνικά δίκτυα. Είναι θέματα για τα οποία πετύχαμε συμβιβασμό. Έχουμε επίσης συνένεση όσον αφορά τον στόχο του 10%. Είναι σημαντικό να γίνουν τα βήματα για καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των χωρών και να πετύχουμε κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Χρειαζόμαστε όμως και τους συμπληρωματικούς περιφερειακούς στόχους. που διευκρινίζουν καλύτερα το τι θα χρειαστεί στο μέλλον, ποια είναι τα σημεία συμφόρησης τα οποία θα πρέπει να εξαλείψουμε. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε τι είδους επενδύσεις χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Απομένει μια κρεμότητα. Δεν έχουμε πιστεί απόλυτα ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Έχει να κάνει με τον ε, συνδυασμό, με, με, με, με τους δεσμευτικούς στόχους, binding targets. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Κύπρος χρειάζεται πολύ μεγάλες επενδύσεις για να πετύχει το στόχο του 10%. Εάν έχουμε δεσμευτικούς στόχους, υποχρεωτικούς στόχους, αυτή η ήπια προσέγγιση που είχαμε μέχρι τώρα όσον αφορά τον στόχο του 10% δεν ε, θα μπορεί να ε, συνεχιστεί, διότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Μετά έχουμε την Ιβυρική Χερσόνησο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Ιβυρική Χερσόνησος ε, δεν έχει 10% ε, διασύνδεση. Χρειάζεται περισσότερη διασύνδεση με την ε, Γαλλία και το υπόλοιπο της Ευρώπης. Εάν όμως είχαμε δεσμευτικούς στόχους για κάθε χώρα, τότε η Ισπανία και η Πορτογαλία πληρούν το κριτήριο αυτό, διότι έχουν 10% μεταξύ τους. Οπότε θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς γιατί να επενδύσουμε άλλα χρήματα εκεί. Το ίδιο ισχύει για τι χώρες τη βαλτική ε, Εστονία, Λιθουανία, Λετωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλό ο στόχος του 10%. Χρειαζόμαστε όμως συμπληρωματικού στόχους σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι μπορούμε να έχουμε περιφερειακούς στόχου, για παράδειγμα για την Ιβυρική Χερσόνησο, τη Βαλτική, τη Βόρεια Θάλασσα, και θα μπορέσουμε έτσι να επενδύσουμε τα χρήματα εκεί όπου θα ωφελήσουν περισσότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Τέσσερις από τους οχτώ σκιώδεις εισηγητές άκουσαν την παρέμβασή σας. αγαπητές συνάδελφοι, θα τους δώσω λοιπόν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Έριξεν, για την ε, έκθεση αυτή, η οποία αποτελεί πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας. Ως σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ, ε, εκτιμώ τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε και συμφωνώ με τον Πίτερ όσον αφορά τις παρατηρήσεις του για ε, την ε, κοινή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από το ΕΛΚ ε, για τις παρατηρήσεις τους που μας έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε καλές τροπολογίες. Θα ήθελα να τονίσω κάποιες πτυχές της έκθεσης αυτής στο όνομα της ομάδας μου. Πρώτον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η παραγωγή ενέργειας είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτή η βασική αρχή, κατά τη γνώμη μου, δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο σχέδιο έκθεσης και γι' αυτό έχουμε υποβάλει σχετική τροπολογία. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτόματη σύγκρουση ανάμεσα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και τους ε, στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ενέργεια και το κλίμα. Δεύτερον, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στηρίζουμε το στόχο του 10% όσον αφορά την ε, διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητο να έχουμε στόχους για να έχουμε μια λειτουργική και ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Έχουμε κάποια νησιά ενεργειακά στη Βαλτική και αλλού στην Ευρώπη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια τροφοδότησης και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Είναι όμως και σημαντικό ο στόχο του 10% να μην είναι αυτός ο σκοπός. Ε, θα πρέπει η έκθεση να αντικατοπτρίζει και τη ε, δυνατότητα πρόσβαση ε, στις υπάρχουσες υποδομές, άσχετα από το αν πληρείται ο στόχος του 10% ή όχι. Επίσης, ε, η υποδομή έχει νόημα μόνο όταν χρησιμοποιείται, οπότε ε, προτείνουμε να προσθεθεί και αυτό στην έκθεση. Επίσης, ε, προτείνουμε να έχουμε κατά νου κάποιες σημαντικές παραμέτρους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να διασυνδεθεί με τρόπο βέλτιστο για, ώστε να ωφελήσει τους καταναλωτές και θα πρέπει να συζητήσουμε και την χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που μας παρέχει η Ευρώπη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. E Από το S&D, κύριε Καπισόν. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρε της Επιτροπής και την Επιτροπή για την εισαγωγή. Αυτό θα πρέπει να είναι το ε, πνεύμα της έκθεσης. Γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, ενιαία εσωτερική αγορά και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Γι' αυτό η συγητής τονίζει ότι θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε τη διασύνδεση. Η βασική στόχη της έκθεσης θα πρέπει να είναι ο επικομιτικός διάλογος διαρκής και μόνιμος. Σήμερα όμως δεν είμαι απολύτως ικανοποιημένη από το περιεχόμενο γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν με έχει ικανοποιήσει η ουσία και πώς να με ικανοποιήσει άλλωστε. Έχει χαθεί ο στόχος, ο κοινός μας, ο στόχος που είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Δεν έχω ξεκαθαρίσει τι ζητάει σε όλη την Ευρώπη αναπτύσσονται οι ανανεώσιμες και θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν και σε τιμές προσιτές για τους καταναλωτές. Αυτά είναι οι βασικοί στόχοι που οικειώνται το ελάχιστο του 10% διασύνδεση. Επαναλαμβάνω αυτό θα πρέπει να είναι το ελάχιστο. Η έκθεση το αμφισβητεί και δεν έχει το στόχο αυτό. Γι' αυτό παρακαλώ όλες τις πολιτικές ομάδες να προβληματιστούν και σας ζητώ την απαραίτητη αλληλεγγύη για να προσπαθήσουμε να ποντάρουμε σε αυτό τον κοινό στόχο. Και παρακαλώ να μην αφισβητείτε αυτή την σκοπιμότητα του 10% και να σπάσουν αυτά τα ενεργειακά νησιά, ενεργειακές νησίδες, δηλαδή απομονωμένες περιφέρειες. Αφήστε δε που τα στοιχεία που δίνονται δεν είναι ακριβή. Στην Ιβερική Χερσόνησο δεν ισχύει το 10%, ούτε 3 με 4% δεν έχουμε και μέχρι το 2020 δεν πρόκειται να έχουμε φτάσει στο 10% με τα σημερινά στοιχεία. Παρακαλώ λοιπόν να δείξετε αλληλεγγύη. Ξέρω ότι και από τις άλλες πολιτικές ομάδες ε, οι συνάδελφοι ε, προέρχονται από χώρες όπου είναι πολύ μεγαλύτερη η διασύνδεση και ίσως δεν έχω καταφέρει να τους πείσω ότι εμείς προερχόμαστε από περιφέρειες που είναι όντως ενεργειακές νησίδες και δεν έχουν την απαραίτητη ε, διασύνδεση. Ακόμα και ο κύριος Κανιέτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμεσα επανέλαβε τη δέσμευσή του να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και να προχωρήσουμε σε διασύνδεση. Και να είναι ένα ελάχιστο το 10% για να υπάρχει μια ουσιαστική και γνήσια εσωτερική αγορά ενέργειας. Ευχαριστώ. Ε, thank you, Ευχαριστώ, κύριε μου. Κύριε Στελίσκα. Καλησπέρα σας. Ξέρω ότι είναι ήθιστε να ευχαριστούμε πάντα τον εισηγητή, αλλά το κάνω πολύ ειλικρινά, γιατί ήταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί του και εκτιμώ επίσης ε, την συμβολή των άλλων συναδέλφων σκιωδών εισηγητών. Εγώ θα είμαι λίγο περισσότερο πολιτικός στην παρατηρήσή μου. Ο στόχος δεν είναι νέος, θα θυμάστε το 2002 ήδη ο στόχος αυτός υπήρχε. Εργαζόμαστε με αυτό το στόχο και ξέρουμε ποια είναι η ισχύουσα κατάσταση 13 χρόνια μετά δεν είμαστε σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε, να διορθώσουμε, να φτιάξουμε σωστά την έκθεσή μας, να εντοπίσουμε τα πραγματικά ζητήματα, της ε, τα σημεία συμφόρησης, αλλά και να ε, θέσουμε στόχους που να είναι ε, διαχειρίσιμοι. Δεν θα ήθελα το 2020 ή το 2025 να φτιάξουμε ακόμα μια έκθεση που θα επαναλαμβάνει το περιεχόμενο ετούτης εδώ. Το σχέδιο είναι νομίζω αρκετά καλά ισορροπημένο και θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω σημαντικές διαφορές ή δυσκολίες ίσως περισσότερο, όσο περισσότερο χρόνο ε, το μελετάμε τόσο περισσότερες τροπολογίες ε, δεχόμαστε και κάπως έτσι ε, αποδυναμώνεται το κείμενο ενώ θα θέλα να είναι πολύ πιο στιβαρό το μήνυμα και να σταλεί μηνύματα επικοινωνιακά πολύ συγκεκριμένα και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μην μπαίνουν ε, σε αυτό το παιχνίδι των τροπολογιών γιατί τελικά όπως σας είπα αποδυναμώνει το κείμενο. Θα κάνω ένα σημαντικό σχόλιο, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να παραμελούμε την, να αγνοούμε την αγορά. Όλοι οι συνάδελφοι που μίλησαν, μίλησαν για την αγορά του ηλεκτρισμού, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και να σεβαστούμε ποιες είναι οι ροές, οι ενεργειακές ροές, οι ροές ηλεκτρικού, ηλεκτρισμού, ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθμίζουμε τις διασυνδέσεις που είναι λυπήσεις αλλά δεν θα πρέπει να κατασκευάσουμε κάτι το οποίο δεν θα αντιστοιχεί στις ροές της αγοράς. Αυτό νομίζω μέχρι στιγμή το έχουμε σωστά πετύχει στην έκθεση. Ίσως να υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις ε, και ίσως κάποιοι συνάδελφοι να μην είναι πολύ ικανοποιημένοι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε επίσης εδώ είναι να βασιστούμε σε αποδείξεις, σε μαρτυρίες, σε πραγματικά στοιχεία δηλαδή, τον αντίκτυπο επιπτώσεων και αυτό επίσης πιστεύω ότι σωστά αναφέρεται εδώ. Ο συνάδελφος, από το Σοσιαλιστές μίλησε για αλληλεγγύη και εγώ αυτό βεβαίως το συνυπογράφω, αλλά θα έλεγα ότι πρόκειται για αλληλεγγύη και υπευθυνότητα και όσον με αφορά εξ ονόματος της Άλτε, εγώ δεν το βλέπω το θέμα από εθνική πλευρά, ίσως κάποιες χώρες να είναι σε διαφορετική θέση. Εγώ εξετάζω το θέμα άσχετα από τις χώρες και τις ε, περιφέρειες, αλλά σκεφτόμενος ε, τους βασικούς στόχους. Πιστεύω λοιπόν ότι το ζήτημα της Ιβυρικής Χερσονήσου θα μπορέσει να εξεταστεί, αλλά θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσαμε να έχουμε μια καθολική προσέγγιση και να ε, εξετάσουμε ίσως ε, και από περιφερειακή άποψης το θέμα. Αλλά μην επικρατήσει αυτή στην έκθεση. Μια-δύο παρατηρήσεις. Νομίζω ότι το εξή σημείο αντικατοπτρίζεται και στο έγγραφο, ελαφρώς πιο αποδυναμωμένο και σίγουρα δεν θα θέλω να αποδυναμωθεί περαιτέρω. Πάντως, δεν θα πρέπει να δαπανάτε ενέργεια και χρήματα μόνο για, τις, για τα πλέγματα αλλά θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και για τις επενδύσεις σε εθνικά δίκτυα. Χρειάζεται αυτή η ισορροπία γιατί διαφορετικά θα κατασπαταληθούν χρήματα και είμαι ευτυχή που η εισηγητή το έχει πλήρω λάβει αυτό υπόψη. Τελευταία μου παρατήρηση αφορά τη δεσμευτική φύση των ποσοστώσεων. Προσωπικά εγώ είμαι ανοιχτό γι' αυτό. Αλλά πιστεύω πως ο εισηγητής έχει δίκιο όταν λέει ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που τουλάχιστον είναι αντιφατικά και εδώ θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Τέλος, εάν θέλουμε να δούμε ε, περιοφέρειες όπως η Βαλτική, αναφέρθηκε και η Βυρική Χερσόνησος, αλλά θα πρέπει και η Βαλτική να εξεταστεί. Θα πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό και να σκεφτούμε και τη σταδιακή μορφή του εγχειρήματο. Πάντως, εν γέννη, Πρόεδρε, πιστεύω πώ είμαστε στη σωστή πορεία. Συμφωνώ με τον εισηγητή πω αν είμαστε κάπω ε, πειθαρχημένοι με τι τροπολογίε ε, θα τα καταφέρουμε και σύντομα. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι εδώ και λίγο καιρό και εισηγήτρια για την εν λόγω έκθεση και πρέπει να σας πω ότι ο εισηγητής έχει ε, ε, βάλει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία στην έκθεσή του, βέβαια πάντα σε συνεργασία με τους σκιώδεις. Πολύ ωραίο αυτό που λέει για την περιφερειακή διάσταση και το φωτίζει πολύ καλά, αλλά και για τη διασύνδεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και ο ρόλος του ΕΙΣΕ, που θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ε, ως προς ανθρώπινους αλλά και τους οικονομικούς πόρους, είναι πολύ σημαντικό και στα θέματα του δικτύου. Υπάρχει μια διασύνδεση που είναι πολύ καλή Αυστρίας, Γερμανίας και λειτουργεί πολύ καλά και αυτή αμφισβητείται πάντα και από τον ίδιο τον συντονιστή των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, τον Acer. Για ποιο λόγο. Στην έκθεση θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο και στην ανάγκη διαφοροποίησης, πιστεύω, των πηγών ε, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα την ενεργειακή ασφάλεια, όπως είπε το πρωί και ο Επίτροπος Άριας Κανιέτε. Και στα πλαίσια της Ενεργειακής Ένωσης το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Αυτό είναι για μένα σημαντικό, ίσως μπορούμε να το τονίσουμε ακόμα περισσότερο και το ίδιο αφορά και τη χρηματοδότηση που μπορεί κάπως ακροθυγός να το ε, εξετάζει η έκθεση, αλλά είναι πολύ περίπλοκο γιατί ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τις γραμμές ε, ηλεκτρικής ενέργειας είναι 52 έργα προτεραιότητας, υπάρχουν οι πηγές πολύ συγκεκριμένες, στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προσεχώς, σήμερα το Connect Europe, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και τα διαρθρωτικά προγράμματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Όλα αυτά δεν χρειάζεται να παραμείνουμε σε γενικότητες. Και ε, για μένα έχει σημασία να μιλήσουμε και για την αδειοδότηση. Γίνεται λόγος για 3,5 ε, χρόνια, αυτή είναι η επιταχυμένη διαδικασία, το fast track ε, για προγράμματα γενικού συμφέροντος. Και στη δική μου τη χώρα, την Αυστρία, η αρκεία της αδειοδότησης είναι πολύ μεγάλη. Και δεν δημιουργούνται πολλές υποδομές. Αυτός ο στόχος του 10% ε, με βρίσκει σύμφωνη και θα το διατηρούσα και θα το έβαζα όμως ε, ελάχιστο στόχο. Όποιος ε, είναι υψηλότερο στη διασύνδεση, σήμερα υπάρχουν κράτη-μέλη, Καλώ, αλλά το 10% να είναι το ελάχιστο. Το είπε και συνάδελφο από την Ισπανία. Για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν συζητούμε για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Και ξέρουμε ποιες άλλες μορφές ενέργειας μπορεί να οδηγήσουν στην ε, δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διασύνδεση και ο περιφερειακός χαρακτήρας που ε, αναφέρεται πάρα πολύ καλά. Στην επόμενη συνεδρία των οικειοδών εισηγητών θα τα ξανασυζητήσουμε και είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Έχω άλλους δύο μιλητές κύριος Τζορίνιο και μετά η κυρία Ένς. Δεν ξέρω αν θέλει κανένας άλλος. Uh, please let me know. Now, Ο κύριος Τζορίνιο. Okay. Yes. Yes, okay. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Επίτροπο Αρίας Κανιέτε. Κατέστη αφές ότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές διαστάσεις. Η μία είναι ε, το σχέδιο της ε, αγοράς ενέργειας και έπειτα από την άλλη πλευρά έχουμε τη μορφή διακυβέρνησης αυτού αυτής της αγοράς ενέργειας ε, και συγκεκριμένα το έγγραφο του Συμβουλίου. Αυτό που προβλέπεται είναι η ενισχυμένη συνεργασία. Οι χώρες δηλαδή θα υποβάλουν εθνικά σχέδια και κάθε δύο χρόνια θα γίνεται αξιολόγηση το, της επίτευξης των στόχων. Εάν δεν υπάρχει όμως ένα ε, στιβαρό στη σύστημα διασυνδέσεων που δίνει την σφαιρική διάσταση ε, των 28 χωρών ε, συνδυασμένων θα διαλυθεί το σύστημα θα, θα αποσυντεθεί. Ε, στο, η αγορά της ενέργειας ε, θα αντιμετωπίσει βραχικυκλώματα και γι' αυτό γνωρίζοντας ε, την ε, εργασία που έχει γίνει πιστεύω πως δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση αυτού του προβλήματος δεν υπάρχει μια σφαιρική εικόνα Επίσης περιέχονται ορισμένες προκαταλήψεις όσων δεν έχουν το πρόβλημα της διασύνδεσης και εγώ δεν μιλάω για άλλη αλληλεγγύη, αλλά μιλώ για λογική. Για λογική. Χωρί τι μίνιμουμ διασυνδέσει, ενιαία αγορά ενέργεια δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει στην Ευρώπη. Thank Σας ευχαριστώ, η κυρία Έρνεστ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Ε, Προ το παρόν ακόμα δεν έχω κλωνοποιηθεί. Έχουμε διάφορε συνεδριάσει δεξιά και αριστερά. Τρέχω, αλλά τα κατάφερα να έρθω. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του και ε, για τις, ε, τις συμβαστικές προτάσεις που είναι καλές και έχει συμπεριλάβει πολλά από όσα πρότειναν οι σκιώδεις. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το πρόβλημα και νομίζω η κατεύθυνση που προτείνει ο εισηγητή είναι απολύτω σωστή. Σε ό,τι αφορά το 10% τώρα τη διασύνθεση, από χέρι γνωρίζουμε ε, ότι εμεί δεν ήμασταν ικανοποιημένοι. Τι θα πει 10% 15% αυθαίρετα είναι αυτά τα πράγματα, κολοκυθιά. Και στη διασύνδεση βεβαίω πρέπει να καλυφθεί το κενό αλλά η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα δεν είναι η ίδια. Ορισμένοι το έχουν καταφέρει αυτό και το ξεπέρασαν κατά πολύ και το αποτελεσματικό και το αποφασιστικό ερώτημα μάλλον δεν είναι η διασύνδεση αλλά να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην αγορά ενέργειας. Και επίσης να ποντάρουμε και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο καθένας μπορεί να συζητήσει ε, μαζί μας ό,τι θέλετε για τη διασύνδεση, αλλά θέλουμε να εστιάσουμε στις ανανεώσιμες, να μην λαμβάνονται απλώς γενικό υπόψη, αλλά να προτιμούνται και να προωθούνται. Ε, ε, για το Acer τώρα, την αρχή αυτή συντονισμού των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, στη δική μας πολιτική ομάδα αυτό το όργανο είναι αμφιλεγόμενο. Δεν ξέρω, κατά πλειοψηφία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί για τους γνωστούς λόγους που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Νομίζω και εγώ ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο εργαλείο, αλλά ε, πρέπει να σας πω κιόλα ότι στην πολιτική μας ομάδα χρειάζεται συζήτηση, δεν το έχουμε συμφωνήσει ακόμα. Όχι εγώ δηλαδή. Ε, κάτι που δεν μας ικανοποιεί και το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι αυτό ε, από τις βόρειες χώρες είναι οι ε, ιστορίες ε, με ε, παραγωγή ενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα. Τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε ξανασυζητήσει και από πλευράς περιβάλλοντος και για άλλα όλες αυτά τα αιωλικά πάρκα και ανεμογενείς μέσα στο πέλαγος είναι θέματα που δεν μας ικανοποιούν. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορούμε να το συμφωνήσουμε και όπως έχει διατυπωθεί στην έκθεση. Για την Ισπανία επίσης έχουμε επιφυλάξεις για το κατά πόσο πηγαίνουν τα πράγματα τόσο καλά όσο λέτε. Δεν είμαι απολύτως βέβαιη, θα το συζητήσουμε όμως και με τους Ισπανούς μας ε, συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ισπανούς συναδέλφους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Κόφουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την ενδιαφέρουσα και πολύ καλή έκθεσή του. να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Σωρίνιο. Πέρα από τον σχεδιασμό της αγοράς και την δομή της διακυβέρνησης, νομίζω ότι είναι πολύ ε, σημαντικό να έχουμε σαφή ευρωπαϊκή πρόπτικη. Το συζητήσαμε αυτό νωρίτερα και με τον Επίτροπο Κανιέτε. Ο στόχος του 10% θα πρέπει να εξεταστεί ε, μαζί με τα εργαλεία. Ε, θέλουμε ολοκλήρωση του δικτύου και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις κοινέ πολιτικές, αλλά ε, και ε, τα, τους διάφορους οργανισμούς ε, όπως την Acer. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη διασύνδεση. Θα πρέπει να τονίσουμε τα εργαλεία και να έχουμε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την έλλειψη διασύνδεσης. Επίσης νομίζω ότι ακόμα έχουμε κάποια σημεία συμφόρησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Είναι ντροπή ότι μιλάμε για την ενιαία αγορά, ε, αλλά δεν την έχουμε επειδή έχουμε αυτά τα σημεία συμφόρησης που δεν έχουμε καταφέρουμε να εξαλείψουμε. Τέλος. Όταν μιλάμε για το δυναμικό της αγοράς, επειδή θέλουμε να αλλάξουμε την ε, ενέργεια μας να γίνουμε πιο ε, βιώσιμοι και να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, τις διασυνδέσεις αυτές. Ευχαριστώ όμως τον εισηγητή για την ενδιαφέρουσα έκθεση και προσλέπω στη συνέχιση των συνομιλιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει. Η ενίσχυση της ενεργειακής υποδομής είναι ένα από τα στοιχεία κλειδί για να πετύχουμε την ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας. Χρειαζόμαστε καλύτερη διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε όμως μόνο στον στόχο του 10%. Γι' αυτό συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, αλλά και τις πηγές στα διάφορα κράτη-μέλη, καθώς και την ποιότητα των εθνικών δικτύων. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να σκεφτούμε ότι κάποιες ελλείψεις στο γερμανικό δίκτυο ε, μπορεί να είναι εις βάρος των δικτύων των γειτονικών χωρών. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα εθνικά δίκτυα. Σημαντικό στοιχείο για να πετύχουμε τον στόχο αυτόν θα είναι να εξαλείψουμε τα σημεία συμφόρησης και να πετύχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών πολιτικών χρησιμοποιώντας ε, χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα μας επιτρέψει να μεταφέρουμε την ενέργεια εκεί όπου την έχουμε περισσότερο ανάγκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κλέιζερ, παρακαλώ. Συγγνώμη που δεν προφέρω σωστά το όνομά σας, είπε ο Πρόεδρος. Από τη Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια ισορπμένη κατά τη γνώμη μας έκθεση. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι ο στόχος της ελάχιστης ε, ε, διασύνδεσης ε, ύψους 10% και τονίζω το ελάχιστης έχει να κάνει όχι μόνο με την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, έχει να κάνει και με την ε, τροφοδοτική ασφάλεια καθώς και με την ενίσχυση ε, της βιωσιμότητας μέσω του δικτύου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι ισορροπημένη η προσέγγιση αυτή και πιστεύουμε ότι με, τους μη με τον μη δεσμευτικό στόχο η έκθεση αυτή ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ευελιξία που δεν αποκλείει την αλληλεγγύη, που δίνει όμως μεγαλύτερο περιθώριο για να ληφθούν υπόψη οι εθνικές και περιφερειακές διαφορές. Όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης, με βάση τον ε, κατάλογο των ε, έργων κοινού ενδιαφέροντος, των PCI, ε, διαπιστώνουμε ότι μεγάλο πρόβλημα είναι η αποδοχή του κόσμου. Θα πρέπει να, να σέβονται τα κράτη-μέλη το χρονοδιάγραμμα των 3,5 ετών και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσουν τη σωστή υποδομή ώστε οι ανάδοχοι των έργων να μπορέσουν να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να δημιουργήσουν υποδομές που να πληρούν ε, την προδιαγραφή αυτή των 3,5 ετών. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τα έργα κοινωνικού ενδιαφέροντος, αλλά και για άλλα έργα στις ε, εγχώριες αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Θα παρακαλέσω τώρα τον εισηγητή να ξαναπάρει το λόγο για να κλείσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις τους. Και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ευρεία πλειοψηφία για να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά αυτά κοινά προβλήματα. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ σε κάποια κοινά προβλήματα της Ευρώπης. Ας ξεκινήσω από την πατρίδα μου. Έχουμε καλή διασύνδεση ανάμεσα στη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, και την Πολωνία, Σουηδία και Γερμανία, αλλά δεν είναι πάντα ανοιχτές οι δίωδοι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η διασύνδεση δεν είναι πάντα το πρόβλημα, πρέπει ε, να είναι και ανοιχτή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αρχές αρμόδιες για την σωστή λειτουργία του συστήματος. Ε, άλλο πρόβλημα Έχουμε με την Πολωνία. Κύριε Πρόεδρε, εσείς προέρχεστε από την Πολωνία. Και η Πολωνία κατά κάποιο τρόπο είναι ενεργειακό νησί, έχει ελάχιστε διασυνδέσεις με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε εδώ λοιπόν περισσότερες διασυνδέσεις. Τρίτο πρόβλημα διαπιστώνεται στη Γερμανία, ανάμεσα στο βορρά και στο νότο της Γερμανίας. Στην περίπτωση αυτή ο στόχος του 10% δεν θα αποτελέσει λύση. Είναι σημαντικό να λυθεί το πρόβλημα ανάμεσα στην Βόρεια και την Νότια Γερμανία. Εάν λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα λυθούν και πολλά άλλα προβλήματα διασύνδεσης ε, στην κοινή αγορά, όπως για παράδειγμα με την Πολωνία. Τέταρτο πρόβλημα είναι αυτό της Ιβηρικής Χερσονήσου, που είναι πολύ λίγο συνδεδεμένη με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Αυτό είναι περιφερειακό πρόβλημα και ο, ακόμα και δεσμευτικός ο στόχος ε, για το 10% αναχώρα δεν θα λύσει το πρόβλημα, ενώ εάν έχουμε περιφερειακούς στόχους θα καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό και πιστεύω ότι ήταν πολύ καλός ο στόχος του 10%. Θα είναι καλό να συνεχίσουμε με τον στόχο αυτό, ενδεχομένως με στόχο 15% μέχρι το 2030, αλλά χρειαζόμαστε μια συμπληρωματική θέση για το, θέμα αυτό. Στην κυρία Ernst, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι το θέμα της διασύνδεσης αφορά όχι μόνο την κοινή αγορά, έχει να κάνει και με τους στόχους για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η κοινή αγορά ευνοεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 80% των, ε, του θέματος των επενδύσεων ε, για τη διασύνδεση συνδέεται με τις επενδύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερη διασύνδεση λοιπόν θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους που αφορούν την αλλαγή του κλίματος ε, Έτσι λοιπόν και στο Παρίσι θα είναι καλό ε, να πετύχουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, έχουμε λίγα λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν να πω κάτι. Δεν αναφερθήκατε στις χώρες της Βαλτικής. Είπατε ότι είναι ενεργειακό νησί, αλλά είναι πολύ καλά συνδεδεμένες με την Ρωσία. Είναι συγχρονισμένες οι χώρες αυτές με τη Ρωσία και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν επαρκεί διασυνδέσει. Ε, για παρατήρηση κάνω, διότι αναφέρατε πολλά ενεργειακά νησιά εντό εισαγωγικών, αλλά οι χώρε τη Βαλτική είναι με σημαντικό πρόβλημα. Ο εισηγητή. Ο λόγο που δεν το ανέφερα είναι ότι πολύ σύντομα θα λυθεί μεγάλο μέρος αυτού του προβλήματος ε, το Νοέμβριο. Θα ε, τεθεί σε λειτουργία νέα διασύνδεση ανάμεσα στη Σουηδία και τη Λιθουανία. Και στο πολύ εγγύς μέλλον προβλέπεται διασύνδεση των βαλτικών χωρών ε, με την Πολωνία. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις αυτές, γιατί είναι πολύ σημαντικές για όλους μας. Η κυρία Κάπεσον Λουίς. Να εκμεταλλευτώ το ότι υπάρχει ακόμα λίγο χρόνος. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω πως έχουμε δίκιο γιατί βλέπω ότι και άλλοι συνάδελφοι το είπαν το ίδιο. Το σχέδιο αυτό άκουσα από την Κομισιόν να λέει ότι είναι ισορροπημένο γιατί επιτρέπει την αλληλεγγύη ώστε να επιτευχθεί αυτό το 10%. Όμως αυτή, αυτός ο εθελοντισμός που υπάρχει εδώ είναι κάπως πεπαλαιωμένος. Η αλληλεγγύη πρέπει να μπει εδώ σε αυτή την έκθεση αλλά πιστεύω πως χρειαζόμαστε εγγυήσεις και συγκεκριμένα στοιχεία για να δώσουμε κίνητρα στην, ε, στον τομέα της ενέργειας. Όπως και εσύ, λέγατε και εσείς, ε, Πρόεδρε, είναι το θέμα του το, το περιφερειακό, του περιφερειακού στόχου. Εφόσον δεν έχουμε 10% διασυνδέσεις, είναι πιθανόν να μην το πετύχουμε αυτό το 10%. Διασυνδέσεις με το η Πορτογαλία, ας πούμε, έχουμε και πάνω από το 10% αλλά δεν είναι αρκετέ για να εγγυηθούμε την ε, ενεργειακή αλληλεγγύη ε, ούτε φτάνει για να μπορέσουμε να ε, δώσουμε ανανεώσιμη ενέργεια. Να καθησυχώσω εδώ και την κυρία, να εδώ και την εκπρόσωπο της ΓΟΕ για την Ισπανία ότι δουλεύουμε πολύ με τους, τις ανανεώσιμες πηγές Βεβαίως ε, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ε, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα σε μια δύσκολη κατάσταση ε, και ιδιαίτερα για την Ισπανία, αλλά αυτό δεν έχει σχέση και δεν σημαίνει ότι η αγορά της Ισπανίας στις ανανεώσιμες πηγές δεν είναι βασική. Έχετε δίκιο ότι είναι σημαντική και για τη Βαλτική και όχι μόνο για την Ιβηρική Χερσόνησο και ελπίζω πως θα συνεχιστεί αυτός ο επικοδομητικός διάλογος για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ευαισθησίες. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη Πρόεδρε που δεν ήμουν εδώ από την αρχή για λόγους ε, εργασίας αλλά όπως επειδή είμαι δραστήρια σε αυτό το θέμα μέσω των τροπολογιών που είναι το βασικό μας έργο των Ευρωβουλευτών που δεν είμαστε ούτε σκιώδεις ούτε εισηγητές. Θέλω να επιμείνω στα όσα είπε η συνάδελφος Καμπεσόν, η συνάδελφος από τους σοσιαλιστές σε σχέση με την Ισπανία και θέλω να πω και κάτι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις διασυνδέσεις. Η δυνατότητα, η ανανεώσιμε πηγέ να συνεχίσουν να αναπτύσσονται όπω μέχρι τώρα στην Ισπανία έχει μεγάλη σχέση με την υλοποίηση των διασυνδέσεων, διότι οι διασυνδέσει θα διευκολύνουν σε συγκεκριμένε στιγμές όταν υπάρχουν ε, πλεονάσματα παραγωγή όπως τώρα με τις ανανεώσιμε, να υπάρχει δυνατότητα να διοχετευτεί αυτή η ενέργεια μέχρι έξω από την Ισπανία μέσω αυτών των διασυνδέσεων. Γι' αυτό και είναι σημαντικέ οι διασυνδέσει, γιατί η διασύνδεση α πούμε, με την Ισπανία γίνεται μέσω τη Γαλλία. Δεν υπάρχει αντίφαση εδώ. Θα πρέπει να υπάρχει θετική σύνδεση ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί ο σημαντικός ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Όπως βλέπετε, είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο και μπορούμε, ε, με το που έχουμε λίγο χρόνο, να προσθέτουμε και να συζητάμε συνέχεια. Να προσθέσω επίσης ότι στην περίπτωση των ανανεώσιμων πηγών έχουμε διάφορα ε, πλάνα στα διάφορα οπότε είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός. το να ανοίξει η αγορά για την ανανεώσιμη, τον ανανεώσιμο ηλεκτρισμό αμέσως τώρα και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για μας τώρα γιατί ο ανταγωνισμός, ανοιχτή αγορά, ε, εμπόριο θα γινόταν με τελείως διαφορετικά σχέδια. Γι' αυτό και είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Για να σταματήσει λοιπόν για να σταματήσουν ε, τα κίνητρα, οι επιδοτήσεις για οποιαδήποτε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να είναι απαραίτητο, ίσως αρχίζοντας από το 2020. Όπως είπα πριν από τρεις ώρες, μαζί με τον Επίτροπο Κανιάτε. Εγώ κάτι τέτοιο πρότεινα. Το 2020 λοιπόν να αρχίσουμε ένα ελεύθερο εμπόριο τότε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Σιγητά ή ίσως η Επιτροπή, έχουμε ακόμα 6 λεπτά. Δεν είναι απαραίτητο να πάρετε το λόγο για 6 λεπτά, όχι, δεν μην σας ορίζω. Στο τέλος της συζήτησης προέκυψε κάτι σημαντικό, σημαντικό θέμα ε, είναι να βελτιωθεί το σύστημα διασυνδέσεων και να ενισχύει η διασύνδεση γιατί έχουμε μεγάλο δυναμικό στις ανανεώσιμες πηγές. Έχουμε στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική Θάλασσα, έχουμε πολύ καλό δυναμικό στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη αλλά και στην Ιβηρική Χερσόνησο. Εάν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα της, της αγωγής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους χρειαζόμαστε περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια και πρέπει να ανοίξει το, το δυναμικό να ελευθερωθεί το δυναμικό αυτών των πηγών στην ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύω πως στο μέλλον το σύστημα ηλεκτρισμού θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο, θα καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι του ενεργειακού συστήματος και αυτό είναι πολύ καλό διότι τα ορυκτά καύσιμα, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Εάν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον ηλεκτρισμό και το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούμε να λύσουμε πολλά από τα μεγάλα μας προβλήματα για την ενέργεια και να πετύχουμε και τους κλιματικούς στόχους, αλλά και την επάρκεια με δική μας παραγωγή, αντί να εισάγουμε από ανατολικές πηγές. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, η ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης έχει προβληθεί για τη 13η Οκτωβρίου ενεστώτος έτους στην Επιτροπή μας και αργότερα στην Ολομέλη. Και πάμε στο επόμενο σημείο υπαριθμό 15, ε, αποστολή της Ήτρες στη Δανία 18-19 Ιουνίου 2015. Ενημέρωση. Είχαμε υψηλού επίπεδο εκπροσώπηση And, uh, the... και επικεφαλής ήταν ο συνάδελφος Μόρταν Χέλβεκ Πέτερσον, αντιπρόεδρος και πρέπει να πω ότι μεταξύ άλλων η αποστολή διερεύνησε το τι κάνει η ε, Κοπενχάγη ε, για να είναι ο ως προς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2025. Και επίσης ε, μας ενδιέφεραν επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά κέντρα, τη βιομηχανία κτλ. Και ε, γενικά έχετε μια αναφορά ε, στο φάκελό σας, γραπτή έκθεση ε, των πεπραγμένων, αλλά να ακούσουμε τον επικεφαλής να μας τα πει και ο ίδιος αντιπρόεδρος κύριος Πέτερσον. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ εξαιρετική η αποστολή αυτή. Στο πρόγραμμά μας είχαμε πολλά από τα κεντρικά θέματα της Επιτροπής μας. Όπως πολύ σας αναφέρατε, επισκεφτήκαμε την Κοπενχάγη και συζητήσαμε της ευφυής πόλης, ε, την ε, προσέγγιση των πόλεων ε, στην δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης. Η Κοπεχάγη έχει την φιλοδοξία μέχρι το 2025 να είναι πόλη ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και Συζητήσαμε τους τρόπους να επιτεθούν φιλόδοξοι στόχοι όπως είναι αυτός. Επίσης, ε, επισκεφτήκαμε την Ένωση Βιομηχανιών της Δανίας ε, και συνομιλήσαμε με πολλές ε, επιχειρήσεις που καταναλώνουν πολύ ενέργεια. Ακούσαμε για παράδειγμα από μια εταιρεία παραγωγής τσιμέντου τι προσπαθεί να πετύχει εξοικονομώντας ενέργεια ενώ είναι ταυτόχρονα μια επιχείρηση ε, υψηλή κατανάλωση ενέργεια που προσπαθεί να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Ε, Επίση ακούσαμε ε, επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και δεδομένου ότι επισκεφτήκαμε και κάποιες επιχειρήσεις ε, ανεμογεννητριών ε, και ανανεώσιμων πηγών ε, ενέργειας. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Επίσης επισκεφτήκαμε την Novo Nordisk που είναι φαρμακευτική εταιρεία. Επισκεφτήκαμε το χημικό της εργαστήριο και συζητήσαμε συζητήσαμε τα πειράματα σε ζώα, σε ζώντα ζώα. Επίσης επισκεφτήκαμε την Green Lighthouse. Επισκεφτήκαμε την Velux, την Danfoss ε, και εξετάσαμε τις δικές τους ε, προτάσεις για επίτευξη της ουδετερότητας ως προς το διοξίδιο του άνθρακα. Και τέλος, ε, επισκεφτήκαμε παράκτιο αιωλικό πάρκο. Ε, επισκεφτήκαμε το μεγαλύτερο του είδους του στη Δανία που ε, παράγει 400 ΜΒ ε, ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε 400.000 νοικοκυρά της Δανίας. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μόνο το μέγεθος και η κλίμακα αυτού του εγχειρήματος ε, ήταν ενδιαφέρον. Αυτό βρίσκεται όχι στην ε, Βαλτική, αλλά στο Σκάγερα και βόρεια του νησιού Ζήλαντ, στον δρόμο προς την Νορβηγία. Είναι τεράστιο το έργο αυτό και ήταν ε, ενδιαφέρον υπό το φως των συζητήσεων που έχουμε στην Επιτροπή μας, που συζητάμε πότε θα γίνει ανταγωνιστική η ενέργεια και από εμπορικής πλευράς. Την ε, μέρα της άφηξής μας είχαμε εκλογές ε, στην Δανία και γι' αυτό πολλοί πολιτικοί ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι με άλλα πράγματα και δεν είχαν καιρό να ασχοληθούν μαζί μας. Ε, δεν μπορεί όμως κανείς να το προγραμματίσει αυτό. Αυτό λίγο μας δυσκόλεψε, αλλά Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει ε, με ανθρώπου στη Δανία. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία και, τα... και του ευρωβουλευτέ που συμμετείχαν. Ήταν ε, μεγάλο προνόμιο η επίσκεψη αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την γραμματεία για την διοργάνωση. Ήταν μεγάλη χαρά και πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανείς να προσθέσει κάτι. Δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Νομίζω ότι ακούσαμε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το θέμα αυτό. Το επόμενο θέμα μας είναι η ενημέρωση σχετικά με τους εξελίξει τριμερείς διαλόγους. Καταρχάς έχουμε τον ε, Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Ο ε, συνάδελφος Σον Κέλλη δεν είναι παρόν, δεν μπόρεσε να προεδρευτεί στις Βρυξέλλες. Προβλήματα με την πτήση του δεν ξέρουμε. Λόγοι υγείας. Ε, ελπίζουμε να είναι υγιής πάντως. Έχουμε άλλους συναδέλφους εδώ όμως και πολύ σημαντικά θέματα. Δίκτυο και ασφάλεια των πληροφοριών. Οδηγία. Η κυρία Πιλάρτε Καστήλο Βέρα. Ξεκίνησε τις εργασίες της ως εισηγήτρια και σχεδόν τις έχει ολοκληρώσει πάνω στην οδηγία αυτή. Η, η Ήτρε είναι επιτροπή που νομοθετεί σύμφωνα με το άρθρο 54. Δεν ήμασταν όλοι παρόντες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας ε, που έγινε η ψηφοφορία και το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την πρώτη ανάγνωση τον Μάρτιο του 2014. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις τον Οκτώβριο του 2014 στην αρχή της θητείας μας δηλαδή. Είχαμε τέσσερις τρίμερις διαλόγους και η συνάδελφός μας θα μας πει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές που δώσατε. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω λοιπόν δεν χρειάζεται δηλαδή να σα εξηγήσω πότε είναι η πρώτη ψηφοφορία κτλ. Τα είπατε εσεί, όπω και εσεί αναφέρατε, ξεκινήσαμε τους τριμερεί διαλόγου ε, τον Οκτώβριο του 2014. Ο τελευταίο τριμερή διάλογο έγινε πριν τι θερινέ διακοπέ ε, στι 20 Ιουνίου του 2015, Φέτο δηλαδή. Είμαι βέβαιη ότι το γνωρίζετε όλοι. Να σας θυμίσω όμως ότι ο στόχος αυτού του σχεδίου οδηγίας είναι να διασφαλίσει την κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει τα κράτη-μέλη και οι φορείς των ζωτικών υποδομών να μπορούν να αντιμετωπίσουν κυβερνοεπιθέσεις. Αναφέρατε και την συμμετοχή της Ήτρη, η οποία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού. Η αρμόδια επί της επιτροπή είναι η ΙΜΚΟ. Η ΙΤΡΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στο θέμα ε, στο θέμα των ε, ομάδων ε, έκτακτης παρέμβασης για τους υπολογιστές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίζουν κάθε κρίσιμος τομέας που καλύπτεται από την οδηγία να έχει μια τέτοια ομάδα έκτακτης επέμβασης και να μπορεί η ομάδα αυτή να χειριστεί ε, τα σχετικά περιστατικά. Επίσης δημιουργείται δίκτυο μεταξύ των ομάδων αυτών ε, με, μέσα, εντός του οποίου γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και εξετάζονται ιδέες όπως είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ποια είναι τα βασικά θέματα που μπορεί να ενδιαφέρουν την Ήτρε. Υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητές της. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο θέλει να είναι πιο φιλόδοξη η συνεργασία εντός του δικτύου ΣΕΡΤ, των ομάδων αυτών δηλαδή. Πράγματι, ε, στην πρόταση η συνεργασία αυτή είναι προαιρετική σε μεγάλο βαθμό. Έτσι λοιπόν δεν είναι πια υποχρεωτική η συνεργασία. Έτσι κινδυνεύουμε η συνεργασία αυτή τελικά να μην είναι πολύ αποτελεσματική. Γι' αυτό θέλουμε πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Από την άλλη μεριά πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με το αν το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας θα πρέπει να διευρυνθεί για να καλύπτει όχι μόνο τις ζωτικέ υποδομές, τις κρίσιμες υποδομές. Έχουμε εδώ γενικά τέσσερις τομείς. Παροχή νερού, ενέργειας, οι μεταφορές ε, και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί τομείς. Τώρα όμως συζητάμε τη δυνατότητα στην πρόταση της Επιτροπής να συμπεριλάβουμε και τις υπηρεσίες της ε, ε, κοινωνίας ε, της πληροφορίας. Εάν συμπεριληφθούν και αυτές οι υπηρεσίες, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις προτείναμε οι υπηρεσίες αυτές να θεωρηθούν όχι οι κρίσιμες ε, ζωτική σημασία υποδομές, αλλά βασικές υποδομές ε, και να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει πρόληψη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αλλά η προστασία σε σχέση με το επίπεδο της προστασίας των χρήσιμων υποδομών, των ζωτικών υποδομών, ε, να είναι κάπως πιο χαμηλό. Το θέμα αυτό εκκρεμεί ακόμα και δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για τον επόμενο τριμερή διάλογο, μάλλον όμως θα πραγματοποιηθεί. Ε, αρχές Δεκεμβρίου θα σας ενημερώσουν. Στο μεταξύ, αν έχει κανείς ερωτήσεις, ευχαριστώ να σας απαντήσω και διμερός Θα χαρώ να μοιραστώ μαζί σας οποιαδήποτε πληροφορίες ή σκέψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πιλά. Και μετά το διμερή διάλογο που θα ακολουθήσει θα μας αναφέρετε ξανά εσείς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Σκιώδη ηγητές δεν έχουμε, γιατί έχει τελειώσει. Ε, κατά την περασμένη θητεία υπόθεση αυτή έχει ολοκληρωθεί από εμά, οπότε οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν ορίσει σκιώδης. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μία πρόταση σχεδίου οδηγίας το Φεβρουάριο του 2013, δηλαδή πριν από δυόμιση χρόνια. Εάν εγκριθεί θα είναι ε, το πρώτο οριζόντιο εγκάρσιο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Δηλαδή είναι ιστορικό αυτό. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, οργανωθεί και όλα τα κράτη-μέλη για να καταπολεμήσει ε, τα προβλήματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου. για τις προτάσεις σας. Θα δούμε ενδεχομένω πώ χρειαστεί και άλλη προσεχή οδηγία στο μέλλον. Είναι πολύ νωρί και πολύ δύσκολο μιλήσει για την επόμενη οδηγία πριν ολοκληρωθεί ο ε, ημερή διάλογο για την παρούσα. Είναι μεγάλε οι δυναμίε και τα προβλήματα και τα αναφέρατε και εσεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τον χρόνο σα και για τον κόπο σα και για τα όσα μα είπατε. Και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι λύσεις διαλειτουργικότητας ε, και συνεργασίες για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, ε, Εταιρείες και πολίτες ως μέσο εξυγχρονισμού του δημοσίου τομέα. See, ε, Και όπως βλέπετε, η ψηφιακή ένωση η ψηφιακή ένωση λέγω είναι πολύ σημαντική εξίσου με την ενεργειακή ένωση ε, την παρούσα θητεία και είναι καινοφανή αυτή η πρόταση γιατί την περασμένη φορά είχαμε πει ότι ό,τι είχε να κάνει με την ενέργεια ήταν πιο σημαντικό και τα ψηφιακά και όλα αυτά. Τώρα η ψηφιακή ένωση είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα ή το θεματολόγιο μα. Ο συνάδελφος μα λοιπόν Κάλλος ε, Σοχίνιου είναι αρμόδιος για αυτό το θέμα, στο πρόγραμμα ΙΣΑ 2 όπως λέγεται, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το τρέχον ΙΣΑ. Σκέτο. Από τον Ιανουάριο του 2016 μάλλον, οπότε δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Ε, διεξήχθη τριμερής διάλογος στις 2 Σεπτεμβρίου. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την απόλυτη μου συμφωνία καταρχήν για τη σημασία της Ενεργειακής Ένωσης και της Ψηφιακής Ένωσης ως δύο μεγάλοι και σπουδαίοι κινητήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περίοδο που ε, βιώνουμε, που ζούμε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έφτασαν στη συμφωνία σε σχέση με το πρόγραμμα ΙΖΑ 2. Είμαστε λοιπόν σε θέση να προχωρήσουμε στη ε, ρυθμιστικά μέσα και θα είναι κανονικά ε, δυνατόν από την 1η Πρώτου 2016 να τεθεί σε πλήρη ισχύ το πρόγραμμα αυτό και να αντικαταστήσει το προηγούμενο που ολοκληρώνεται στα τέλη του 2015. 131 εκατομμύρια ευρώ έχει αυτό το πρόγραμμα για να αναπτυχθούν ε, σε λύσεις ε, ε, διαλειτουργικότητας για τα δημόσια ιδρύματα αλλά και για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Αλλά το πρόγραμμα που προκύπτει δεν είναι απλώς συνέχεια του προηγούμενου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, υπάρχουν δύο κεντρικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα της νέας ενιαίας ψηφιακής αγοράς και κατά δεύτερο λόγο υπήρξε μια τεχνολογική εξέλιξη πολύ μεγάλη τα τελευταία χρόνια. Και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι έχουν γίνει σημαντικές ε, ε, τροπολογίες για τις οποίες ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αγωνίστηκαν και το Συμβούλιο τελικά τα δέχτηκε. Θα σας τα συνοψίσω, θα σας πω τα πιο σημαντικά. Από αυτά τα συστήματα που στην Επιτροπή μας στην Ήτρε, που ήταν ε, η αρμόδια από τις ουσίες, είχαμε την ΙΝΚΟΜ, της Τρίγης Αγοράς και τη Λίμπε των πολιτικών ελευθεριών. Τα θέματά μας, από τα θέματά μας λοιπόν καταφέραμε κάτι το οποίο θεωρούμε πως είναι καθοριστικό, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό να μην ε, στηρίξει απλά μόνο λύσεις ιδιαλειτουργικότητας, μάλιστα δεν θα υποστηρίξει κυρίως ε, λύσεις διαλειτουργικότητας, αλλά θα υποστηρίξει επίσης κοινέ πλατφόρμες, κοινέ βάσεις, κοινέ γλώσσες, κοινά εργαλεία, θεμέλια επί των οποίων ε, οι διάφορες διάφοροι διοικητικοί μηχανισμοί θα μπορέσουν να στηρίξουν τις λύσεις τους. Είμαστε δηλαδή σε ένα επίπεδο πριν από το επίπεδο των λύσεων των ίδιων. Αλλά μπορούμε αυτά τα 131 μα εκατομμύρια να ε, πολλαπλασιάσουμε πολύ περισσότερο τις δυνατότητες των διοικητικών μηχανισμών και να να αυξήσουμε τον ε, τις συναλλαγές και τις ανταλλαγές, την διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε αυτές. Επίσης έχουμε βάλει ε, τρεις ε, ε, στόχους, τρία κριτήρια για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων. Κυρίως μιλήσαμε για την, την εδαφική κάλυψη. Στα παλιότερα προγράμματα γινόταν χρηματοδότηση κυρίως εθνικών λύσεων, ενώ τώρα ε, έχουμε δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ε, εδαφική κάλυψη. Επίσης αξιοποιήσαμε ε, το γεγονός ότι οι λύσεις αυτές θα πρέπει να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν στις νέες πλατφόρμες και επίσης στηρίξαμε πολύ την απλοποίηση των διαδικασιών έτσι ώστε να είναι ένα πρόγραμμα πιο εύχριστο. Επίση, καταφέραμε να μπει η αρχή του κινήτρου για την δημιουργία κοινοτήτων χρηστών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία και, και ε, επαφή ανάμεσα στους χρήστες, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τους πολίτες τους τελικούς χρήστες δηλαδή, τους καταναλωτές και ε, τους χρηματοδότες του προγράμματος. Η πιο απλή λύση ήταν να προβλέψουμε τη δυνατότητα να υπάρχει ε, πρόσβαση από πλευρά της κοινωνία των πολιτών. Αυτό δεν ήταν δυνατόν, ήταν όμως δυνατόν να εισαρθεί αυτή η αρχή της δημιουργίας κοινοτήτων που θα αξιολογήσουν online επιγραμμικά στη διάρκεια της ε, ε, ε, προετοιμασίας των προγραμμάτων και να μπορέσουν να προτείνουν βελτιώσεις. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό κέρδος το οποίο ε, ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την εσωτερική αγορά ε, και δίνει, δίνει μεγαλύτερο βάρος στις δημόσιους μηχανισμούς και, την, και τις επιχειρήσεις πολέμηση από την ψηφιακό αποκλεισμό με, πιο, με λύσεις πιο ευνόητες για τους πολίτες και λιγότερο γραφειοκρατικές για τις επιχειρήσεις. Και τέλος, καταφέραμε να βρούμε ένα σημείο επαφή, ένα σημείο ισορροπίας σε σχέση με ένα πολύ σημαντικό θέμα που ήταν ένα θέμα το οποίο ε, απασχόλησε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, δηλαδή η διασφάλιση των κριτηρίων προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικού χώρου ανα πάσα στιγμή της περίοδου εφαρμογή αυτού του προγράμματος που θα ισχύσει ανάμεσα στο 2016 και το 2020 και ξέρουμε ότι ε, αυτοί οι κανόνες προστασίας των δεδομένων είναι, είναι κανόνες και, και, ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη και θα ε, απο, ε, και ε, έγινε δεκτό ότι ανα πάσα στιγμή στην εξέλιξη του προγράμματο θα τηρούνται οι ισχύουσες νομοθεσίες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε πως είναι τελικά καλό αυτό το πρόγραμμα και θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφους για την εξαιρετική του συμμετοχή και τους και οδησυσυγητές, του συναδέλφους από τις άλλες επιτροπές την Ήμικο και τη ΛΥΜΠΕ και επίση όλη την τεχνική ομάδα του Κοινοβουλίου, τις διάφορες υπηρεσίες, τα γραφεία της ε, Κομισιόν και της ε, Επιτροπής. Υπήρξε λοιπόν εξαίρετη συνεργασία σε αυτή την ε, προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Όλα φαίνονται θετικά λοιπόν αυτά που είπατε. Ελπίζω λοιπόν ότι στις 13 Οκτωβρίου θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε τη συμφωνία. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα πρέπει να στέλνει μια επιστολή που επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι, εστάλει, εστάλει. Να περιμένουμε να μας έρθει. Όχι, όχι κύριε Πρόεδρε. Τη λάβαμε αυτή την επιστολή. Λάβαμε την επιβεβαίωση από την Προεδρία. Όλα είναι έτοιμα για την ψηφοφορία. Πολύ ωραία λοιπόν. 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ συνάδελφε που επιτύχατε συμφωνία και που δώσατε τόσο μεγάλη ε, όθηση σε αυτό το ζήτημα. Διάφορα. Σας ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρίαση 12 Οκτωβρίου. Α, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή είμαστε στη συζήτηση των διαφορών, τη δυνατότητα από πλευρά της, της Επιτροπής να συνεδριάσουμε εκτάκτως για το ζήτημα που αφορά το πρόβλημα της Volkswagen. Νομίζω πως ε, η Επιτροπή μας είναι αυτή που είναι αρμόδια για τέτοιο είδους ε, ζητήματα που προέκυψαν ε, στη ΣΥΠΑ, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί να προκύψει τέτοιο ζήτημα και εδώ στην Ευρώπη. Γι' αυτό ρωτώ τον Πρόεδρο αν είναι δυνατόν να διοργανωθεί μια έκτακτη συνεδρίαση ad hoc για το πρόβλημα της Volkswagen, που θεωρώ πως είναι πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Ναι, βεβαίω. Ε, καταγράφουμε το έτοιμά σα. Είναι σημαντικό. Μάλλον θα πρέπει να διευρύνουμε το πρόβλημα όχι μόνο για μια ευρωπαϊκή κινητοβιομηχανία, αλλά και στις υπόλοιπες. Γνωρίζουμε ότι το μεταξύ είναι υπό εξέλιξη διαπραγματεύσει TTIP και ότι και ότι αυτές περιλαμβάνουν τέτοια ζητήματα όπως αυτό της Volkswagen ε, στην ΕΠΑ και θα το σκεφτούμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό που ζητάτε. Μάλιστα. Ο κύριος Μαρτένς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σε επιστήσω την προσοχή στο εξής. Σήμερα το πρωί αναβλήθηκαν ε, πολλές ε, ψηφοφορίες για εκθέσεις, είδαμε τι συνέβη το πρωί. Εντάξει, κατανοώ ότι τα λέει ο κανονισμός όλα αυτά, αλλά προσβλέπω στη δική σας βοήθεια και υπολογίζω σε αυτή, έτσι ώστε το συντομότερο να ψηφιστούν αυτές οι εκθέσεις. Διότι είχαν ήδη εγγραφεί για ολομέλειες στο Στρασβούργο, στην ημερήσια διάταξη και δεν θα επιθυμώ τώρα να το παραπέμψουμε αυτό στις καλένδες επειδή δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε επί του κανονισμού ε, προσβλέπω σε εσά για να συγκληθεί ενδεχομένω έκτακτη συνεδρία τη επιτροπή μα στο Στρασβούργο για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Ε, βεβαίως, το κατανοώ αυτό. Ε, δεν θα το παραπέψουμε στι καλένδες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίω θα πρέπει να ψηφιστούν το συντομότερο δυνατό. Οι εκθέσεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εξασφαλίσουμε. Για να μεταφραστούν όλες οι τροπολογίες. Ξέρετε αγαπητέ συνάδελφε, περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να μεταφραστούν όλες οι τροπολογίες. So, yeah, is no, no translation, no, no interpretation now. Έχετε πρόβλημα με τη διερμηνία. Μιλάει για τη μετάφραση ο πρόεδρος. Ε, θα πρέπει να μεταφραστούν όλες οι τροπολογίες. μετάφραση, όχι τη διερμηνία, να μεταφραστούν οι τροπολογίες και ξέρετε ότι στο Λουξεμβούργο είναι οι μεταφραστές μας. So it's quite different issue. Okay, dear friends. Λοιπόν, αυτά. Επόμενη συνεδρία σε 12 Οκτωβρίου το απόγευμα και 13 Οκτωβρίου το πρωί και το απόγευμα ραντεβού σε λίγες εβδομάδες, α και προηγουμένως στο Στρασβούργο φυσικά, όπου ψηφίζουμε στην Ολομέλη. Ευχαριστώ πολύ.